Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Παρακαλώ, καθίστε, διότι όπως γνωρίζετε θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και θέλουμε να μπορείτε να ακούσετε υπό καλές συνθήκες τον Επίτροπο. Όπως γνωρίζετε, ο Επίτροπος Σαστιλιανίδης χθες το βράδυ επέστρεψε από την Δυτική Αφρική, όπου μαζί με τον Επίτροπο Ανδρουκαΐτη εξέτασαν την κατάσταση όσον αφορά τον ιό έμπολα επιτόπου. Ο Επίτροπος παραβρέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι η πρώτη του δημόσια ε, δήλωση σχετικά με αυτά που είδε, αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να μάθουμε από τη Δυτική Αφρική, από την κατάσταση στη Δυτική Αφρική. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι θέλουμε να σας στηρίξουμε ε, με οποιονδήποτε τρόπο για να ελέγξουμε την επιδημία. Έχουμε και τον εισηγητή μας τον κύριο Γκόενς, ο οποίος εκπονεί έκθεση πρωτοβουλίας για τον ιό έμπολα και τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες του. Προτού να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, μπορούμε παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημέρησια διάταξη. Συμφωνείτε όλοι. Ούτως ή άλλως μόνο ένα θέμα έχουμε στην ημέρησια διάταξη. Μου λένε όσον αφορά την διερμηνία λόγω της ε, συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό, ε, που είναι πολύ σημαντικό θέμα και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν έχουμε διερμηνία στα κροατικά, ρουμανικά και τσέχικα. Και πορτογαλικά παρέχονται μόνο παθητικά. Μπορείτε να μιλήσετε, όχι όμως να ακούσετε, διότι όπως ξέρετε συγκαλέσαμε τη συνεδρίαση πολύ αργά, διότι συμφώνησε ο Επίτροπος να έρθει αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Δυτική Αφρική. Κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο για να μας περιγράψετε τις εμπειρίες σας από τη Δυτική Αφρική. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Προτού να αναφερθώ στον ιό έμπολα, επέτρεψέ μου να πω, επίτρεψέ μου να πω πόσο ε, έχω συγκλονιστεί από, τον, από τη δολοφονία του Πίτερ Κάσινγκ. Είναι μια πράξη βαρβαρότητας η οποία υπογραμμίζει πόσο ε, επικίνδυνη είναι η ζωή των ανθρώπων που, εργάζονται, που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να τον τιμήσω και όσους δολοφονήθηκαν πριν από αυτόν από το Ισλαμικό κράτος. Πραγματικά είναι απίστευτο το γεγονός αυτό. στις 30 Σεπτεμβρίου δεσμεύτηκα μπροστά στην Επιτροπή σας. Η πρώτη μου επιστολή, αποστολή συγγνώμη, ως Επίτροπος να είναι προς τις χώρες που ε, έχουν πληγεί από τον ιό έμπολα. Χθες επέστρεψα από μια τετραήμερη επίσκεψη στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης αποστολής. Ήταν συγκλονιστική η εμπειρία μας. Είδαμε από πρώτο χέρι, επί τόπου, τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Νιώσαμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ενώ σε κάποιες περιοχές φαίνεται να υποχωρεί η νόσος, σε άλλες δυστυχώς εξαπλώνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Γενικά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον φόβο να υπαγορεύσει τις ενέργειές μας. Η προσέγγιση μου ήταν σαφής από την αρχή. Θέλουμε να αποκλείσουμε, να απομονώσουμε τον ιό, όχι τους ανθρώπους στις χώρες που έχουν πληγεί. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σύνθημα, πιστεύω η νόσος έχει επηρεάσει αρνητικά την κοινωνία στις χώρες αυτές. Έχει καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό. Έχει τραυματίσει ανθρώπους. Η διαδικασία ανάκαμψης θα είναι δύσκολη και θα απαιτήσει πολύ χρόνο. Γι' αυτό η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μακροπρόθεσμη. Διασφαλίζω τους ανθρώπους στις τρεις αυτές χώρες ότι δεν αγωνίζονται μόνοι τους ενάντια στον ιό έμπολα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι θεωρητική, είναι απτή. Επιτρέψτε μου δύο πράγματα. Καταρχάς, να σας παρουσιάσω την εικόνα της κατάστασης όπως την είδα εγώ στις χώρες αυτές και δεύτερον, να τονίσω τους πιο βασικούς τομείς όπου προτίθεμε να αναλάβω δράση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η αποστολή μας είχε δύο στόχους. Καταρχάς, να στείλει ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η Ευρώπη είναι παρούσα, ότι πρέπει να νικηθεί ο ιός κυρίως στις χώρες αυτές και δεύτερον να εντοπίσουμε τα βασικά κενά στην αντίδρασή μας, να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, τώρα πια είναι πολύ ουσιαστική. Επιτόπου είδα τη συγκεκριμένη δουλειά που ε, κάνουν πολλά κράτη-μέλη μας. Στη Γουινέα μέρος του προγραμματός μου ήταν κοινή επίσκεψη ε, με τον Υπουργό ανάπτυξης της Γαλλίας Ανίκ και χάρηκα που είδα πώς εντείνει η Γαλλία τον ρόλο της εκεί. Στη Σιέρα Λεόνε είδα την εξαιρετική δουλειά που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και είδα πολλά παραδείγματα του πώς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν ζωτική βοήθεια. Επίσης, συνάντησα ε, ε, ανθρώπους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και ε, ντόπιου και ε, από διεθνείς οργανισμούς και ενθάρρυνα τις θαρελές προσπάθειές τους και διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν στιγματίζονται από τις κοινωνίες τους όταν επιστρέφουν από τις αποστολές τους. Χρειάζονται λοιπόν την υποστήριξή μας. Επιπλέον, ε, συνάντησα επιζώντες του ιού έμπολα. Οι προσωπικές τους ιστορίες είναι συγκλονιστικές. στα μάτια τους. Μπορούσε κανείς να δει τη χαρά τους που είναι ακόμα ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα και τον πόνο τους που έχουν στιγματιστεί και έχουν τεθεί στο περιθώριο από μέλη των οικογενειών τους και των κοινοτήτων τους. Πολλοί από αυτούς τώρα είναι εθελοντές ε, στην προσπάθεια να σώσουν τις ζωές άλλων. Και οι επιζώντες λοιπόν χρειάζονται την μακροπρόθεσμη βοήθειά μας, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό τομέα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι εξή. Αυτά πρέπει να κάνουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ένα βασικό συμπέρασμα λοιπόν είναι να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες. Η επιδημία έχει αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο στις τρεις αυτές χώρες. Όπως ε, και έχει διαφοροποιηθεί η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Συνεπώς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις προσπάθειές μας. Καταρχάς, ε, να αναφερθώ στη Σιέρα Λεόνε να ξεκινήσω από τα καλά νέα. Οι επιτόπου δομές για συντονισμό των προσπαθειών ε, είναι ισχυροί. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά συντονίζοντας ε, την πολιτική και στρατιωτική προσπάθεια μαζί και με άλλους διεθνείς εταίρους επισκέφτηκα το κέντρο εκπαίδευσης ε, που διαχειρίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Είδα την εξαιρετική δουλειά που κάνει η ομάδα του Ηνωμένου Βασιλεία, του Βασιλείου όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου, την ανοικοδόμηση τοπικού δυναμικού και ε, όσον αφορά τη διοχέτευση των πόρων εκεί όπου ε, είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Επίσης, ε, συνάντησα τον πρόεδρο Κουρούμα και την ε, κυβέρνησή του και είναι η ισχυρή μου εντύπωση ότι ε, επικεντρώνουν τις, τους, τις προσπάθειές τους. Τώρα όσον αφορά τα λιγότερα καλά νέα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών στη Σιέρα Λεόνε. Σε μερικές περιοχές δυστυχώς η αύξηση είναι δραματική χρειάζεται, απαιτείται περισσότερο γιατρικό προσωπικό και περισσότερα κέντρα περίθαλψης. Όχι σε τρεις εβδομάδες, τώρα. Πρόκειται σαφώς για έναν τομέα όπου μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα. Σε στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο για να διαπιστώσουμε πού είναι πιο σημαντικές οι ανάγκες. Το ERCC της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διατεθειμένο να βοηθήσει και είναι έτοιμο από κάθε άποψη. Δεύτερον, Λιβερία. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ενθαρρυντικά στοιχεία ο αριθμός των περιστατικών φαίνεται ότι σταθεροποιείται σε κάποιες περιοχές της Λιβερίας, όπως και στην Σιέρα Λεόνε. Είναι πολύ ισχυρή πολύ ισχυρές οι δομές επιτόπου. Όλοι οι φορείς συνεργάζονται στενά για να διαπιστώσουν την εξέλιξη της νόσου. οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και πολλά κράτη-μέλη μας κάνουν πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά. Ωστόσο, οι εν μέρη ενθαρρυντικές τάσεις της προηγούμενης εβδομάδας δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν να ε, υποτιμήσουμε την κατάσταση. Στη Λιβερία, πιθανότατα να βλέπουμε πιο γρήγορη μεταφορά της νόσου και θα πρέπει να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντικό δυναμικό σε κάποια κέντρα περίθαλψης. Επισκεφτήκαμε ένα από τα κέντρα αυτά έξω από την Μονρόβια, αλλά χρειαζόμαστε μικρότερες ομάδες άμεσης αντίδρασης. Κάτι που τόνισε και η πρόεδρος Τζόνσον Σίρλιφ. Τέλος, Γουινέα. Εδώ η εικόνα είναι περίπλοκη. Ενώ παραμένει πολύ πιο χαμηλός ο αριθμός των περιστατικών από ό,τι σε γειτονικέ χώρες, βλέπουμε μια ε, βραδία αύξηση και τα περιστατικά είναι σκορπισμένα σε μεγάλη περιοχή. Επίσης, είναι πιο πολύπλοκη εικόνα όσον αφορά το συντονισμό. απομένει να γίνει πολλή δουλειά για να συντονιστούν οι διάφοροι φορείς, για να έχουμε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της επιδημίας. Χαίρομαι που ο κύριος Ζιραρτάν ε, πρότεινε η Γαλλία να αναλάβει ε, ρόλο ηγετικό. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο Κόντε και θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειες μας επί τόπου. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν κέντρα περίθαλψης, χρειαζόμαστε όμως και μεγάλο αριθμό ανθρώπων που να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Το βασικό πρόβλημα ε, παραμένουν οι τοπικές κοινότητες ε, στα δάση. Για τη Γουινέα λοιπόν χρειαζόμαστε και επιδημιολόγους εκτός από τις ομάδες περίθαλψης και οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι ε, κινητές για να προλαβαίνουν ε, την όσο στα διάφορα μέρη. Υπάρχουν και κάποια οριζόντια θέματα. Καταρχάς, πρέπει να ξεκινήσουν οι προσπάθειες ανοικοδόμησης ε, των συστημάτων υγείας των χωρών αυτών. Εδώ ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να, να συμβάλλουν σημαντικά. Επίσης, συμβολή για το σύστημα MEDEVAC, το οποίο έχουμε δημιουργήσει και το οποίο ενισχύεται περαιτέρω από κράτη-μέλη όπως είναι το Λουξεμβούργο. Τρίτον, ανάγκη για πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της περιοχής αυτής πάνω στον ιό έμπολα. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη η περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση του ιού έμπολα, διότι το πιο επικίνδυνο μέρος είναι ε, εκεί που διασταυρώνουν τα σύνορα των τριών αυτών χωρών. Και βέβαια ενδιαφέρουσα είναι και η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πάνω στα εμβόλια και στην ετοιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για μένα μαζί με τον συνάδελφό μου τον Επίτροπο Ανδρικοαϊτής να επισκεφτώ την περιοχή αυτή. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι για εξάπλωση στην ευρύτερη περιοχή, στο Μάλι για παράδειγμα, μετά από τις πολύ ανησυχητικές περιπτώσεις ε, που είχαμε εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο ε, το σημάδι αυτό. Ποια θα είναι τα επόμενα μου βήματα ως συντονιστής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ιό έμπολα. Οι άμεσες προτεραιότητες μου είναι καταρχάς να δώσω συνέχεια στα ευρήματα της αποστολής αυτής. Ε, να εκπονήσω ένα κατάλογο των όσων απαιτούνται. Απαιτούνται ομάδες περίθαλψης, επιδημιολόγοι, ε, κινητές ομάδες. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την ε, άμεση κινητοποίηση. Το ERCC είναι διατεθειμένο να τα κάνει αυτά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να συγχαρώ τη Σουηδία που ήταν το πρώτο κράτος μέλος που πρόσφερε ε, γιατρική ομάδα στο ERCC. Επίσης, ε, προτείνω να ε, συγκληθεί μια συνάντηση υψηλού επίπεδου πάνω στον ιό έμπολα. Προτείνω να εξετάσουμε την επιδημία σε δύο φάσεις. Καταρχάς, βραχυπρόθεσμα να, να, να αποφασίσουμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας σε συνεργασία με τους άλλους βασικούς παράγοντες και χρειαζόμαστε βέβαια και τη δική σας συμβολή σε αυτήν την διάσκεψη υψηλού επίπεδου που θα γίνει. Και επίσης, μία ευρεία διάσκεψη μαζί με τις χώρες της περιοχής που να εξετάσει επίσης τι θα γίνει μετά ε, τον ιό έμπολα. Από τότε που ανέλαβα ε, τα καθήκοντά μου, Έχω στενή συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους, με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών ε, Εξωτερικής Εδράσης και επίσης με άλλους παράγοντες και γι' αυτό ε, θα φροντίσω το Σώμα των Επιτρόπων να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θα συνεχίσω τη στενή συνεργασία με τα, άλλα κράτη, με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις δράσεις μας και θα σας κρατώ ενήμερους, όπως άλλωστε κάνω και σήμερα, ώστε να μπορώ να ακούσω και τις δικές σας αντιδράσεις. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό που μου είπε ο Ιμπραχήμ, που είναι ένας από τους ανθρώπους στο Κονάκρι που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μου είπε ότι ο ιός έμπολα είναι ευφυής. Αλλά εμείς μπορούμε να είμαστε πιο ευφυείς. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ιμπραχήμ σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αποτίσω φορό τιμή σε όλους τους εθελοντές που είναι επιτόπου και κινδυνεύοντας τη ζωή τους προσπαθούν να σώσουν τις ζωές των άλλων ενώ συγχρόνως είναι εκπατρισμένοι και πολλές φορές επικρίνουν και οι δικοί τους άνθρωποι. Εγώ είχα μία συνάντηση με εκπροσώπους ε, ε, διαφόρων οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού και μου έκαναν αυτή την παρατηρήση. Επίσης, σε αυτούς, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει δεσμευτεί για να καταπολεμήσει τον έμπολα, καθώς και εκπροσώπους των κυβερνήσεων, σε όλους όσους ε, ε, ασχολούνται και με τη διοικητική υποστήριξη και όσους μπορούν ε, να συνεισφέρουν από τι αφορά τη μισή, είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε ευφιέστεροι από τον ίδιο τον ιό. Με άλλα λόγια, εγώ λέω πιο ταχύς, διότι μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι είμαστε πιο αργοί και ίσως κάπως πιο ανόητοι. Θα το λέω ίσως με ομό τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον έμπολα αν είμαστε πιο ευφύς και πιο ταχύς, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα μια καταγραφή των αναγκών. Των αναγκών σε άνδρες, σε γυναίκες, σε υλικό, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη μέθοδο. Και θα ήθελα να κάνω διαφοροποίηση μεταξύ συντονισμού και συντονιστού. Χαιρετίζω όπως όλοι οι παρόντες στην αίθουσα το γεγονός ότι εσείς οριστήκατε ως συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμήσουμε τον έμπολα. Αυτό το οποίο όμως με σοκάρει στον ορισμό σας δεν, είναι, δεν είστε εσείς, αλλά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Πρέπει να πω ότι εκπροσωπεί κράτη-μέλη κάποια τα οποία ε, δεν ε, αντέδρασαν καθόλου και τώρα ζητείτε να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα ο συντονισμός δεν δούλεψε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε εσείς με αποφασιστικότητα να επιβάλλετε την απόψή σας. Εσείς πρέπει να πείτε ποιες είναι οι ανάγκες που έχετε σε προσωπικό, σε υλικό, να πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, να πείτε ποιος θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και σε συνεννόηση και με τους άλλους ε, παράγοντες, παράγοντες τους εμπλεκόμενους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Θέλουμε βεβαίως εμείς να μας πείτε τι χρειάζεστε. Κάθε φορά να μας λέτε τι ακριβώς χρειάζεστε. Πράγμα το οποίο δεν το ξέρουμε προς το παρόν ποιες είναι οι ελλείψεις και επίσης Εάν αποτύχουν οι προσπάθειες κατά του έμπολα εξαιτίας έλλειψης χρημάτων, θα το στιγματίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι μπορούμε εμείς να ε, υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε αποφασιστικότητα στις κυβερνήσεις ότι πρέπει να ενεργήσουν πιο δυναμικά. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αφήσουμε τα πράγματα να επιδεινώθουν. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε ικανότητες μεταφοράς και εκένωσης σε περίπτωση προβλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα master plan στην διάθεσή μας, το περιμένουμε από και ελπίζω ότι αυτή η ικανότητα που θα πρέπει να αναπτύξουμε θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ε, έχουμε περισσότερο προσωπικό επιτόπου. Μετά από τον ορισμό των δικών σας, ε, είπατε ότι θα πρέπει εσείς να πάτε για να δώσετε το πράγμα και ως ιατρός και στους συναδέλφους σας, τους άλλους ιατρούς, ε, για να πάνε επίσης, να ενεργήσουν επίσης. Αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα και σας θαυμάζουμε για αυτό που κάνατε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στην, ε, τον ε, απολογισμό που θα κάνετε, το τι ακριβώς έχουμε, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία εάν επιβρανδυνθεί η οποιαδήποτε διαδικασία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Αναμένουμε λοιπόν από εσάς που να γνωρίσουν οι πάντες ότι εσείς είστε ο καπετάνιος σε αυτή την υπόθεση. Εσείς είστε στην ε, κορυφή της πυραμίδας και ότι πείτε θα πρέπει οι άλλοι ως τη βάση να το εφαρμόσουν και εσείς θα πρέπει να μας πείτε ποιος δεν είναι έτοιμος και διατεθειμένος να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία μας ε, υπαγορεύετε εσείς με τον ορισμό σας ως υπεύθυνο. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά την κινητοποίηση, σε φάση επίγουσας ανάγκης, δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τρομερές λεπτομέρειες θα πρέπει να στοχεύουμε πιο ψηλά από αυτά που χρειάζεται. Θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί από αυτό το οποίο υπαγορεύουν οι σημερινές καταστάσεις. Και είμαστε οι τελευταίοι που θα σας κάνουμε το οποιοδήποτε παράπονο ή θα σας προσάψουμε κάτι αν ζητήσετε περισσότερα κονδύλια από αυτά που χρειάζεστε για να μπορέσετε να κάνετε κάτι επιτόπου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε με ευφύ τρόπο τις ανάγκες, και να μην χάσουμε χρόνο προσπαθώντας να κάνουμε μικρομπακάλικους λογαριασμούς ως το τελευταίο δεκαράκι. Πιστεύω λοιπόν ότι και από αυτής της πλευράς ε, το επίγον της κατάστασης δικαιολογεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μην κάνουμε πραγματικά, επαναλαμβάνω, μπακάλικους λογαριασμούς και ασχολούμαστε με τις δεκάρες. Δεν θα πρέπει αυτό να περιορίσει την δράση μας, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η αριθμητική δεν ε, αξίζει και πολύ. Και βεβαίως ό,τι κάνετε πρέπει να πω ότι είναι ε, κάτι το οποίο υποστηρίζουμε πλήρως. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον Επίτροπο Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Επίτροπο δεδομένου ότι ε, υλοποίησε δύο πολύ σημαντικές υποσχέσεις που μας είχε δώσει. Μας είχε πει ότι η πρώτη του ταξίδι θα είναι στη Δυτική Αφρική, στις χώρες που έχουν πληγεί από τον έμπολα. Δεύτερον, ότι θα επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα την Επιτροπή μας, θα συνεργάζεται στενά μαζί μας και το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ παρόν την ε, επαύριο της επανόδοση από την Αφρική πραγματικά είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερως και το τονίζω. Δύο παρατηρήσεις. Αναφέρατε την ε, συνεισφορά των κρατών μελών. Τονίσατε πώς ενήγησαν κάποιες χώρες και όπως και ο εισηγητής για το έμπολα θα ήθελα να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα όμως να σας κάνω και μια ερώτηση για τον συντονισμό εντός της Επιτροπής και την ε, σχέση που υπάρχει μεταξύ της βοήθειας, της αποκατάστασης και της άπτυξης. Δεδομένου ότι είστε επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά είστε και συντονιστής συγκεκριμένα για τον έμπολα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ίσως θα κάνετε κάποια ταξίδια εσείς ή κάποιος άλλος συναδελφός σας και θα εστιάσετε και στην ε, πολιτική και σε θέματα αναπτυξιακά που πρέπει να ακολουθηθούν και μέσω πρόσφυγμα και μα, μακροπρόθεσμα. Τονίσατε ότι πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσουν τα συστήματα υγείας στις χώρες αυτές να βελτιωθούν, για να μπορούν οι χώρες αυτές να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχαν μέχρι τώρα την ικανότητα να το κάνουν ε, αμέσω μόλις ε, εμφανίστηκε η νόσος αυτή και σε πρώιμο στάδιο. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτησή μου και ένα σχόλιο και τελικά την άποψή σας. Πιστεύω ότι είναι πρωταρχική σημασία, γιατί αναφέρατε ότι είναι πρωταρχική σημασία να, είμαστε, να υπογρυπνούμε συνεχώς. Να ξέρουμε ποιε είναι οι θετικές εξελίσεις, αλλά να είμαστε, να για τα αρνητικά. Όσον αφορά την προσοχή ε, που πρέπει να ε, δώσουν και τα ΜΜΕ και πώς μπορούμε να έχουμε ε, να, να επαγρυπνεί η κοινή γνώμη στην Ευρώπη, να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Ποια είναι μία ε, ισορροπημένη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε να δείτε η σωστή πληροφόρηση και να μην καταληφθεί από φόβο και πανικό ο κόσμος. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ε, ισορροπημένη επικοινωνία. Επίσης, όπως είπαν οι συνάδελφοι, όλες οι πολιτικές ομάδες, όλη η ομάδα πραγματικά σας υποστηρίζει πλήρως σε οτιδήποτε ε, κάνετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δουλειά σας. Πρώτον, τήρησατε το λόγο σας και δεύτερον, στείλατε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, οικοδομήσατε εμπιστοσύνη και κάνατε ορατή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα Καταρχάς να πω ότι πάντα θα πρέπει να τονίζουμε την σημασία των ε, ηρών στην καταπολέμηση του ε, ιού έμπολα, των ανθρώπων που ε, που χωρίς μεγάλες χειρονομίες κάνουν την σημαντική δουλειά σε καθημερινό επίπεδο. Ο κίνδυνος είναι, όπως έχει πει ο Μπανκιμούν, ε, οι τρεις ε, πληγήσεις χώρες ε, να αντιμετωπίσουν λοιμό. Και η ερώτησή μου είναι, υπάρχουν συλλογισμοί σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι παρούσα και το Σαββατοκύριακο είχαμε στο Brisbane το G20 ε, οι απαντήσεις στον ιό έπολα ήταν πολύ απογοητευτικές. Ε, εν μέρει υπόθηκε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση. Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν συμμετάσχει πολύ μέχρι τώρα να ε, συμμετάσχουν πιο ενεργά, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερα, αλλά... Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από πλευράς του G20. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ αδύναμη και απογοητευτική απάντηση. Επίσης, συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης, ε, ούτε κάτι τέτοιο υπάρχει. Και νομίζω ότι ο συνάδελφος έχει απόλυτο δίκιο πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα στα συστήματα υγείας για να αντιμετωπίσουμε, για να προλάβουμε τέτοιες επιδημίες. Σε μια ερώτηση για τη Λιβερία. Η Λιβερία ε, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, πριν λίγες μέρες, ε, κάτι που είναι θετικό, αλλά η απόφαση της Αμερικής ε, να στείλει 3.000 ε, στρατιώτες αντί 4.000 μάλλον ήταν βιαστική απόφαση και για τη Σιέρα Λεόνε είπατε ότι έχουμε συνεχώς ε, νέα κρούσματα και ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται εκτός ελέγχου. Επίσης, όσον αφορά το Μάλι, Διαπιστώθηκαν εκεί περίπου τρεις περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την ε, δέσμευσή σας ε, και ελπίζω και στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά. Η Επιτροπή μας και εσείς. Ευχαριστώ. και κυρία Χόιμπουκ μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική σας απόφαση να επισκεφθείτε αμέσως τις χώρες που έχουν πληγεί από το έμπολα. Χρειάζεται μεγάλο θάρρος, το οποίο έχετε και ως γιατρός βέβαια. Και βεβαίως το ότι κάνατε και μία ε, αποστολή ανείχνευσης του ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Πρέπει να πω ότι εμείς αντιδρούμε πολύ αργά σε τέτοιου είδους ε, γενικότερες καταστροφές και θα αναφέρω το φιάσκο μετά από τα προβλήματα και το σεισμό στην ΑΕΤ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση Ίσως ήταν καλύτερο το σκορ μας από ό,τι στο παρελθόν, και, αλλά θα πρέπει να έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξή. Ποια είναι οι ελλείψεις μας, τα προβλήματά μας. Οι δικοί μας ε, υπουργοί στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν για την κρίση του έμπολα να δώσουν ένα ε, ε, ευρώ. Και ο Μπομπ Γκέλντορφ, ο Μπόνο και άλλοι προσπάθησαν επίσης να συγκεντρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για βοήθεια. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να συνεισφέρει, μπορεί μέσω ίντερνετ να το κάνει με πολύ μικρά ποσά, πέντε λιρών. Υπάρχουν πολλά άτομα λοιπόν τα οποία προσπαθούν να ε, βρουν χρήματα. Πάντα υπάρχουν ε, άτομα τα οποία κάνουν ό,τι μπορούν σε διεθνές επίπεδο για να βρουν χρήματα και πολλές φορές με εκπλησιοποιούν πόσο γενναιόδωρα είναι τα άτομα όταν θέλουν να βοηθήσουν κάποιοι. Στην περίπτωση του τσουνάμι θυμάστε πότε ακριβώς γίνει και πάλι. Ε, τελικά ε, κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί για να βρει χρήματα. Ίσως στην Ευρώπη θα έπρεπε όλοι μαζί από κοινού να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουμε αρκετά χρήματα τα οποία έγκαιρα θα φτάσουν στα χέρια μας. Ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε τα χρήματα. Τι δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί που πρέπει εμείς να στείλουμε για να μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε την ασθένεια και να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. Τι χρειαζόμαστε, εργαζόμενους, ε, οι υγειονομικές υπηρεσίες, πιο θαραλέο προσωπικό, νοσηλευτικό, παρανοσηλευτικό, εξοπλισμό. Τι, τι ακριβώς χρειαζόμαστε, δεν ξέρω τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Η κυρία Χόιμποκ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που κάνατε αυτό το ταξίδι. Έχουμε υποτιμήσει τις πρώτες εκκλήσεις ε, των γιατρών στις χώρες αυτές. Είναι λοιπόν ισχυρό μήνυμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το ταξίδι σας στις χώρες αυτές. Από την αρχή της θητείας μου με κυνηγάει ο ε, ιός έμπολα. Έχουμε σημαντικές ελπίδες από τη δουλειά σας, τον ρόλο που έχετε αναλάβει ως συντονιστής. Είναι σημαντικό λοιπόν να συντονιστούν σωστά οι προσπάθειες ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, τα είπε και ο συνάδελφος. Ε, η ερώτησή μου είναι κάπως διαφορετική. Επί τόπου μπορέσατε να αποκτήσετε μια εικόνα της γενικής οικονομικής κατάστασης. Ε, μπορείτε να μας πείτε, διότι ακούστηκε ότι η οικονομία καταραίει, ότι δεν λειτουργούν οι υποδομές ότι θα δούμε να υπάρχει λοιμός και να μην ε, υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Μπορείτε να μας δώσετε εσείς την εικόνα σας, θα με ενδιαφέρει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μωρίς Πόγκα, αντιπρόεδρος, ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σήμερα πολλοί είναι αυτοί που σας συγχαίρουν για την αποστολή που κάνατε στις χώρες που έχουν πληγεί από τον έμπολα. Να προσθέσω εγώ τα συγχαρητήριά μου. Είπατε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου μας είχατε πει πως πρόκειται να μεταβείτε, το πράξατε. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την δέσμευση που καταλάβετε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε στο θέμα των υποδομών που έχουν ε, οργανώσει άλλα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας για το μέλλον, το όραμά σας για το μέλλον, για την ε, υλοποίηση περαιτέρω υποδομών προκειμένου άλλες επιδημίες να μην αναπτυχθούν στις εν λόγω περιοχές. Δεύτερο ερώτηση. Τονίσατε στην παρέμβασή σας ε, πως υπάρχει ένα συντονισμός που γίνεται σε επίπεδο κομισιών. διαβουλευτήκατε με τον ε, Επίτροπο που ασχολείται με θέματα ανάπτυξης, διότι κατά την μου η σχέση μεταξύ ανάπτυξης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ στενή. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Κύριο Γκερέρο και η κυρία Άννη Σάιντε Πιέρικ θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. προημερών είχαμε μια συνεδρίαση σχετικά με τον έμπολα στην Επιτροπή μας. Μας ενημέρωσε ένας γενικός διευθυντής ε, και συμμετείχαν πρέσβεις ορισμένων χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό του έμπολα και τότε ετέθη το θέμα δύο σημαντικών ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα η αναγκαιότητα να αναπτυχθούν να πτυχθεί άμεσα οικονομική πόρη και να δοθεί βοήθεια και κατά δεύτερο λόγο να προφασίσουμε να αποφύγουμε την δαιμονοποίηση και την απομόνωση των κρατών που όχι μόνο υποφέρουν από την επιδημία αλλά χάνουν και οικονομικούς πόρους διότι οι οικονομίες τους έχουν κουραστεί και δεν μπορούν να ε, κάνουν εξαγωγές. Ε, εντάξει, μπορούμε να καταπολύσουμε την έμπολα, αλλά δεν ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τους ε, πολίτες που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια. Τώρα, για την εξέλιξη των ε, έμπολα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταχύτητα και την επιτάχυση. Στην φυσική και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που σταματήσαμε είναι η επιτάχυνση, αλλά δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε την ταχύτητα. Με άλλα λόγια, συνεχίζει να αναπτύσσεται με λιγότερη βία, λιγότερη ταχύτητα, αλλά θα πρέπει να επιβρανθεί. Όχι μόνο η επιτάχυνση, αλλά και η ταχύτητα. Από πλευρά τώρα δική μας, Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, νομίζω πως ε, έγιναν ε, δύο καλά βήματα, πρώτα συντονιστή και μια μεγαλύτερη δέσμευση του τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών ε, για περισσότερα μέσα, ε, ένα, μέχρι ένα δις ευρώ για την καταπολέμηση του έμπολα. Αλλά θα πρέπει να δράξουμε την σημερινή δυνατότητα που μας παρέχεται για να προωθήσουμε μια πιο εντατική και έντονη απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Ε, πρώτα απ' όλα το ότι επίκειται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Ε, γνωρίζω τα συμπεράσματα, τα προκατακτικά που έχουν προετοιμάσει στην ε, μόνιμες αντιπροσωπίες οι οποίες είναι ε, ξεκάθαρες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του έμπολα. Φυσικά γνωρίζω και την επιστολή σας προς τον πρόεδρο της Κομισιόν για τους στόχους και τις προτεραιότητες. Επίσης, κρίνω ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε από αυτές τις μέρες που έχουμε στη διάθεσή μα, προκειμένου στο Συμβούλιο Υπουργών να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, με σαφή πρόταση θεωρώντας ότι και άλλα σημεία του συμπεράσματα των μονίμων αντιπροσώπων αποτελούν έτοιμα ε, προς τον συντονιστή προκειμένου να ενημερώσει το Συμβούλιο και να υποβάλει προτάσεις ε, προς το Συμβούλιο. Κατά δεύτερον λόγο έχουμε την συνεδρίαση ανωτάτου επίπεδου την οποία αναφερθήκατε στην επόμενη συνάντηση υψηλού επίπεδου, την οποία θα ε, ζητούσα και νομίζω πως ε, τόσο εγώ όσο και το σύνολο της Επιτροπής μας ε, θα συμφωνούσε να σταλεί ε, η, έκθεση του συναδέλφου Γκέρνης νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτήν την συνάντηση υψηλού επίπεδου. Τρίτον, έχουμε την σύνοδο της, των χωρών ΑΚΕ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο. Αφρική, Καραβική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συναντηθούμε με πολλούς εκπροσώπους αυτών της Υπήρου και από γειτονικέ τους χώρες που βρίσκονται εν δυνάμει, εν κινδύνο για την εξάπλωση της επιδημίας θα μπορούσαμε λοιπόν να, συζητήσουμε μαζί το θέμα. Επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο περνάει στα ψηλά και θα πρέπει να το εξετάσουμε από πολιτική σκοπιά. Εγώ θα, ε, θα αρνηθώ ότι είπα αυτό που λέω τώρα, αλλά η Ιταλική Προεδρία είχε την κακή τύχη να ε, προεδρεύει στο δεύτερο εξάμεινο, το οποίο είναι πιο σύντομο από το πρώτο εξάμεινο, κατά στιγμή όπου όλα τα όργανα της Ένωσης είχαν αρχίσει να συγκροτούνται, κοινοβούλιο, κομισιόν κλπ. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό για την, Ευρωπαϊκή, ε, την, συγγνώμη, την Ιταλική Προεδρία να ε, δώσει μια όθηση στο ζήτημα του έμπολα και αν όλοι λοιπόν μπορέσουμε να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τέλος ε, να παρατηρήσω όσο είπατε ότι ε, κάποιος, ε, ο Ιμπρέμ είπε ότι το, ο έμπολα είναι ευφυές ε, ευφυής ιός τώρα. Αλλά το πρώτο στο μέλημα της ευφυίας είναι να κατορθώσει να επιβιώσει. Αλλά θα πρέπει λοιπόν σε εκ του να ε, χρησιμοποιήσουμε την ίδια φασιστικότητα με την φασιστικότητα την οποία έχει δείξει ο ιός του έμπολα για την επιβίωσή του και την εξάπλωσή του. Θα ζητήσαμε λοιπόν, να μας δώσετε κάποιες προφορίες, αν είναι διαθέσιμες τώρα, αν τις έχετε αυτές τις προφορίες, για το πώς θα προχωρήσουμε για να ε, αναπτύξουμε περαιτέρω ιατρικό υλικό στα κράτη-μέλη, στα, στα πληγέντα κράτη, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα οι συστήματα υγείας, ε, τα υγειονομικά συστήματα, δίνοντας μια απάντηση δομική και ο κύριος Στή αναφέρθηκε στο ζήτημα πώς θα ε, μεταφέρουμε αυτές τις ε, θέσεις προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και τέλος ε, να συμφωνήσω με τις παρεμβάσεις ε, οι οποίες έγιναν και τις, για τις ευχαριστίες. Σας, να σας ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου που δουλεύετε έντονα και εντατικά και να συμφωνήσω για αυτές τις ε, σφαγές, για αυτούς τους φόνους που δεν τους κάνει κάποιος ιός αλλά άτομα τα οποία πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν με, ε, με άτομα τα οποία ε, προτείνουν αυτές τις λύσεις. Ευχαριστώ. Άννη Σφάιζερ Πίρικ. Παρακαλώ μου πείτε πώς λέγεται το όνομα, πώς πρέπει να προφέρετε το όνομά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όταν ε, ε, έγινε γνωστή η είδηση για τα, το, ε, τον έμπολα στην Αφρική, η Ευρώπη αμέσως ε, φρόντισε να αντιδράσει. Και μία ερώτηση. Δεν θα ήταν καλύτερο όλοι να γνωρίζουμε τα στοιχεία τουλάχιστον μια φορά το μήνα, να ξέρουμε λοιπόν την πρόοδο αυτής της φοβερής νόσου. Τα αναφέρω αυτά διότι αυτή είναι η έκτη συνεδρίαση, μιλάμε για συντονισμό, για ανθρωπιστική βοήθεια, για χρήματα, πώς θα αντιδράσουμε και ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να ακούσουμε από εσά τώρα είναι ένα πρόγραμμα δράσης. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε σε αυτό το έργο σας και όχι μόνο ως κοινοβούλιο αλλά και ε, για, μιλάω για όλα τα κράτη. Εγώ είμαι Ολλανδί και κάθε χώρα φυσικά χρειάζεται να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η απόψή σας, τι θα πρέπει να συμβεί σε κάθε μια χώρα. Μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια, για ιατρική βοήθεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι συχνά στιγματίζονται κάποια πρόσωπα τα οποία ε, ε, επιθυμούν να μεταβούν στις χώρες αυτές και μετά έχουν πρόβλημα ε, άμα την επιστροφή τους. Και τέλος μιλήσαμε για την επιδημιολογία. Μία συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί Κοιτάξτε, άκουσα πολύ κόσμο και ε, θεωρούν ότι έχουν εγκαταλειφθεί στις ε, χώρες τους. Πώς ε, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε χάρη, τα ορφανά, τα παιδιά τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Ευχαριστώ. Maybe I could just ask, just ask, well, Έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε, να συνοψίσω καταρχά σε μια ερώτηση των συναδέρφων που έχει να κάνει με το σχέδιο δράση. Διότι είπατε ότι θα εντοπίσετε τι ανάγκε που υπάρχουν στι χώρε και νομίζω ότι είναι χρήσιμο αυτό που είπε ο κ. Γκόεν και ο Γερέρο, ότι επίκειται το η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παρασχεθούν ε, όλα αυτά. Επίσης επένεσατε τη Σουηδία που είναι η πρώτη χώρα που ε, θα στείλει ομάδα γιατρών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συντονισμού. Πόσες ομάδες χρειάζεστε. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να γνωρίζουμε πότε θα κινητοποιηθούν, διότι ο κύριος Ντέιβα ανέφερε ότι και το κοινό συμβάλλει χρηματικά στον αγώνα κατά του έμπολα. Αλλά ο κόσμος θέλει να γνωρίζει ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να μου πείτε τι γίνεται, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τις πράξεις μας. Επίσης αναφερθήκατε σε μια διάσκεψη κορυφής. Ελπίζουμε στο τέλος, όταν όλα θα τεθούν υπό έλεγχο, να γίνει μια διάσκεψη για να καταπολεμηθούν και τα άλλα προβλήματα, διότι είπατε ότι καταστρέφονται ζωές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου και αυτό το θέμα στους επόμενους μήνες. Ε, πολλές ερωτήσεις σας θέθηκα, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Yes. Allow me to use my mother tongue. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την μητρική μου γλώσσα διότι θα πρέπει να είμαι σαφής, συγκεκριμένος και να εκφράσω και τις βαθιά μου συναισθήματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω κάτι που νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει από το hearing. Ε, και επειδή το νιώθω θα το πω. Όταν έρχομαι σε αυτή την Επιτροπή παίρνω θάρρος και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εθάριση που μου δίνετε. Νιώθω ότι κινούμαστε στην ίδια γραμμή. Μπορεί να έχουμε μικρές διαφορές στις προσεγγίσεις, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ίδια αγωνία για τα πράγματα. Θα ξεκινήσω με βάση τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις σας και ελπίζω να μπορέσω να σας δώσω συνολικά απαντήσεις. Πρώτον, τελικά το ταξίδι είχε τη συμβολική του σημασία και θα σας πω λεπτομέρειες για την αξία αυτής της συμβολικής σημασίας αλλά την ίδια στιγμή είχε και πολύ πρακτική αξία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε και την πρακτική αξία. Μαζί με τον συνάδελφο Αντριουκάητης στο treatment center στη Σιέρα Λεόνε όπου βοηθούσε τμήμα του Αγγλικού στρατού αποφασίσαμε να υποστούμε τη δοκιμασία, όλη τη δοκιμασία το πώς φοράς τη στολή σε όλες τις ζώνες της διαδικασίας μέχρι να φτάσει στο red zone. Σας λέω ότι ως γιατρός πέρασα πολλές φορές τη δοκιμασία να φτάσω στο χειρουργείο. Ε, αυτή η διαδικασία είναι πιο δύσκολη από τη διαδικασία ενός γιατρού που φτάνει στο χειρουργείο. Γιατί το λέω. Για να καταλάβετε τη σημασία των training centers. Τη σημασία να έχουμε ψηλό επίπεδο ανθρώπων, όχι μόνο στο επίπεδο των γιατρών, αλλά στο επίπεδο των hygienist, στο απλό επίπεδο των ανθρώπων που βοηθούν στα πιο απλά πράγματα του ήρωες του γιατρού χωρίς σύνορα, το MSF. Η δουλειά που χρειάζεται είναι μεγάλη, περισσότερη από, όσοι, από ό,τι φανταζόμαστε. Στο treatment center στη Μονρόβια και ευτυχώς βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες εκτός του ότι συναντήσαμε μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο των MSF, το Mobile Lamp, το Mobile Hospital, συναντήσαμε τους survivors Είδαμε και τους ήρωες, τους γιατρούς μαζί με τους hygienists το πώς μπόρεσαν να φτάσουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο συνεργασίας. Και όταν μιλάμε για νοσοκομείο, μη φανταστείτε τα νοσοκομεία που ξέρουμε εδώ. Μιλάμε για τέντες μέσα σε ένα χώρο κυρίως με χώμα κάτω, με υποτυπώδεις συνθήκες νοσοκομείου. Θα μου μείνει αξέχαστη η συνάντηση με μία νεαρή γιατρό από τη Σουηδία και ένα άλλο νεαρό γιατρό από τη Νέα Υόρκη οι οποίοι σας λέω ως γιατρός κουβεντιάζοντας μαζί τους το επίπεδο της εκπαίδευσής τους ήταν πάρα πολύ ψηλό. Μπορούσαν να ήταν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου ή να ήταν στο private sector και να κάνουν πάρα πολλά λεφτά στη ζωή τους αλλά ήταν εκεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με βοήθεια από ανθρώπους με λίγες δυνατότητες να τους βοηθήσουν και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ένα νέο περιστατικό που σώθηκε, ένα νέο survivor, δεν, δεν μπορεί να φανταστείτε τι έγινε σε ολόκληρη την περιοχή. Τα χειροκροτήματα που άκουσαν και έτρεξαν όλοι να τον φέρουν να αποτυπώσει τα finger points πάνω σε έναν τοίχο που είχαμε όλα τα finger points. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτή η νεαρή γιατρό από την Ουψάλα είναι ένα παράδειγμα που πρέπει κάποια στιγμή να τη φέρουμε στις Βρυξέλλες για να δείξουμε τι σημαίνει ανθρωπισμός. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε ακριβώς για να στείλουμε το μήνυμα. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε να στείλουμε το μήνυμα. Νομίζω έτσι θα δείξουμε στην κοινή γνώμη της Ευρώπης για να περιορίσουμε και την ιστερία αλλά και το φόβο. Και αυτό το σκοπό είχε και η επίσκεψη με τον συνάδελφο Αντρίου Κάιτης. Από την άλλη θα πω και μια άλλη εμπειρία που είχαμε στο Ντόγκα Hospital στην Ουινέα με ένα από τους survivors που επειδή έχει στιγματιστεί πλήρως από το χωριό του δεν μπορεί να επιστρέψει είναι εκεί βολουνθία κάθε μέρα έξω από το νοσοκομείο που είναι στημένο το οι υποδομές των γιατρών δικοσύνορα του MSF και μαζί με τον Ιμπραχήμ ο οποίο και αυτό στιγματιστήκε δεν μπορεί να πάει σπίτι του ή στο κονάκρι το μόνο που ήθελα ήταν μια αγκαλιά μόνο μια αγκαλιά είπατε πριν για τα ορφανά και έχετε απόλυτο δίκιο δεν μπορεί να μην αποφασίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βρούμε τον τρόπο με ειδικό κονδύλι για να φτάσει βοήθεια στα ορφανά. Θα είναι σαν να μην υπάρχουμε ως Ευρωπαίοι με συγκεκριμένες αξίες και αρχές. Ο φίλος ο Γκέρενς ήταν αναγκασμένος να φύγει. Μίλησε και ρώτησε πολύ σωστά τι γίνεται με την καταγραφή των αναγκών. Θα πάρω τη μια, μια χώρα ξεχωριστά. Ήταν τρεις μέρες από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. δεν συναντήσαμε μόνο επισήμους και national coordinators, αλλά είδαμε ανθρώπους από όλε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που βοηθούν από όλα τα UN agencies. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και διαφορές στις εκτιμήσεις. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση για να συμφωνήσουν όλοι. Πήραμε διάφορες πληροφορίες. Κάπου υπήρχαν και έντονες διαφωνίες. Κάναμε τρεις-τέσσερις συναντήσεις με όλους αυτούς τους ε, partners και όντω υπήρχε και έντονη συζήτηση ότι ο ένας έλεγε ότι αυτό είναι το πρωτεύον, ο άλλος έλεγε αυτό είναι. Γι' αυτό θέλει προσοχή και ήρθαμε εφοδιασμένοι για να κάνουμε πολλές συζητήσεις και μεταξύ των commissioners αλλά και με τη βοήθεια των εξαιρετικών συναδέλφων που ήταν μαζί μας από, τα κάπινες αλλά και από την ΕΚΟ για να μπορέσουμε όντως αυτά που είδαμε να τα κωδικοποιήσουμε σε πραγματικές ανάγκες. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Να βάλουμε ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το τρίτο. Ό,τι σας αναφέρω τώρα είναι κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Δεν θα είναι η τελική μας ακτίμηση η οποία θα πρέπει να καταγραφεί για να αρχίσουμε όντως το action plan που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ακόμα τρεις-τέσσερις μέρες αυτές τις μέρες για να γίνει η πλήρης αξιολόγηση του τι είδαμε. Ήδη από αύριο ξεκινούμε συναντήσεις με τους, όλους τους commissioner που έχουν άμεση εμπλοκή στο ζήτημα. Με τον κύριο Μίμητσα θα βρεθούμε γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Είναι ο Commissioner ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως να βοηθά σε πολλά επίπεδα. Στην Λιβερία χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα όχι γιατρού. Χρειαζόμαστε στο επίπεδο των hygienist και nurses, νοσοκόμες και υγιεινιστές, hygienist. Στη Λιβερία η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη από τις άλλες περιοχές. Γι' αυτό έχουμε και τη μείωση των περιπτώσεων. Υπάρχει μια άμεση εμπλοκή του Αμερικάνικου στρατού δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό κέντρο συντονισμού. Η κυβέρνηση και φαίνεται να υπάρχει και από πλευράς αντιπολίτευσης μια, ένα κονσένσους και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό το κέντρο συντονισμού δουλεύει πάνω σε ένα πολύ σύγχρονο επίπεδο με data, computers, είναι ένα επίπεδο που μπορεί να πει κάποιο ότι μπορεί να βρεθεί ανάλογο και σε ευρωπαϊκή χώρα. Είναι όντω το πιο ψηλό επίπεδο που αντιμετωπίσαμε αυτό το κέντρο συντονισμού στη Λιβερία. Γι' αυτό στη Λιβερία η κατάσταση είναι ίσως η πιο ελεγχόμενη, αλλά και εκεί πρέπει ακόμη να είμαστε συγκρατημένοι. Πρέπει να μείνουμε on alert. Σιέρα Λεόνε, βέβαια τα προβλήματα στην οικονομία της κάθε χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εάν δεν υπάρξει ένα ανάλογο του σχεδίου Marshall για τις περιοχές και τις τρεις αμέσως μετά που θα περιορίσουμε το κακό δεν νομίζω να υπάρχει εύκολη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ουσιαστικά έχει καταστραφεί όλος, ο ιστός της οικονομίας. Οι υποδομές όσες υπήρχαν, γιατί εξαιτία των εμφυλίων πολέμων, εξαιτία πολλών προβλημάτων, η κατάσταση και πριν δεν ήταν όντως σε καλά πλαίσια. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και καταλαβαίνετε επιδεινώθηκε ακόμα πιο πολύ. Σιέρα Λεόνε. Το πρόβλημα στη Σιέρα Λεόνε είναι ότι ενώ υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς του Προέδρου, δυστυχώς ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές. Γι' αυτό και αποτυπώνεται στην αύξηση των περιστατικών. επιστρέφοντα στη Λιβερία αυτό που τον ίστιγε στη Λιβερία, επειδή συναντήσαμε και ένα-δυο επιδημιολόγους, από την σου Σουηδό, ο οποίο είναι σύμβουλο της Λιβεριανή κυβέρνηση, πρέπει το συντομότερο στη Λιβερία να κατεβούμε στο επίπεδο των community centers. Χρειαζόμαστε πολύ πιο μικρές ομάδες στήριξης στα χωριά, στα villages, στα, στο επίπεδο του community. Το, το επίπεδο το κρατικό είναι ικανοποιητικό. Πρέπει το συντομότερο. Που αντιλαμβάνεστε ότι εδώ χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτον, κυρίως hygienists και nurses και να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο ως community center. Αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να εμπλέξουμε τις ίδιες τις κοινωνίες που να αναλάβουν τον τρόπο να πείσουν στα χωριά ότι οι κηδείες πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο υγιεινής και όχι με έναν τρόπο μέχρι τώρα με βάση το tradition με βάση τις απόψεις και τις αντιλήψεις ότι οι κυρίες πρέπει να γίνονται ε, όπως γινόντουσαν μέχρι τώρα και είχαμε μετάδοση από τα μπέιραλς του ιού εξαιτία του ότι έπλαιναν τον νεκρό, τον φιλούσαν, γίνοντουσαν οι παραδοσιακές κυρίες που γίνονται στην περιοχή. Χρειάζεται δηλαδή και ενημέρωση μεγάλη και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλές γλώσσες. Γι' αυτό πρέπει να εμπλέξουμε, όπως και στις άλλες χώρες, αλλά και στη Λιβερία, τοπικούς παράγοντες γι' αυτό. Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι αποφασισμένη. Στη Σιέρα Λεόνε πάλι υπάρχει πρόβλημα στο επίπεδο των communities, στο επίπεδο να πιστεί η κοινωνία να τηρεί στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα στο επίπεδο του state. Ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές ενός σωστού operational center. Οι Άγγλοι έχουν κάνει καλή δουλειά στα training centers. Κάθε μέρα εκπαιδεύουν καινούριου Hygienists, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερο. Εκείνο που χρειάζεται να στείλουμε εμείς medical personnel είναι ότι χρειάζεται supervision. Κάποιος χρειάζεται αυτές τις δύσκολες διαδικασίες να τις ελέγχει ως γιατρός, ως ειδικό. Το supervision είναι πολύ κρίσιμο και στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόνε. Θέλω εδώ να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχει να εξασφαλίσουμε το κοντρόλ στο περιβόητο red point, το κόκκινο σημείο που συναντιόνται τα σύνορα, το border point μεταξύ των τριών χωρών. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που μεταδίδεται ο ιός. Εκεί έγινε και η μετάδοση από το πρώτο κρούσμα της Γουινέας που στη Σιέρα Λεόνε και επεκτάθηκε. Αυτή είναι η εκτίμηση επιδημιολόγου. Εκεί ουσιαστικά, και θα το πω διότι μιλάμε ειλικρινά, έχουμε τεχνητά σύνορα, artificial porters. Υπάρχουν οικογένειες και από τις δύο πλευρές των σύνορων, οι οποίες μετακινούνται. Υπάρχει ένας ποταμός, ο οποίος απλώς είναι ένα σύνορο. αυτέ οι οικογένειε αντιλαμβάνεστε ότι μετακινούμενες μεταφέρουν και το πρόβλημα. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει αυτό που είπα πριν, regional cooperation. Πρέπει να πιστούν οι κυβερνήσεις από εμά, από τον διεθνή παράγοντα, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνει αυτό το, η συνεργασία που να ξεκινήσει από το επίπεδο των Προέδρων και να φτάσει στα local authorities, ακόμα και σε leaders, αρχηγούς μικρών communities και μικρών σε μέγεθος φυλών. Γιατί στο forest area και στα χωριά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπάρχει πραγματική άσκηση εξουσίας του κράτους, η οποία βέβαια είναι υποτυπώδης ακόμα και στις πρωτεύουσες. Υπάρχει ένα θέμα governance γενικό. Λοιπόν, πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ το Porter Point μεταξύ των τριών και εκεί θα επικεντρωθούμε πολύ. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν ειδικά treatments και training centers σε αυτό το σημείο. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος το ότι είδαμε την, επισκοπήσαμε την κατάσταση on the ground. ότι χρειαζόμαστε συνεχώς medical supplies and medical equipment, νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι το Ολλανδικό πλοίο έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στο δρόμο και θα φτάσει με βοήθεια από 9 διαφορετικά κράτη, μεγάλη βοήθεια σε υλικό και σε ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα για να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούν σωστά τα mobile labs, τα laboratories. Και πάμε στη Γουινέα που είναι μια περισσότερο ειδική περίπτωση από τις άλλες. Είναι γνωστό ότι στη Γουινέα είχαμε και τα προβλήματα μια resistance απέναντι στο ότι ο έμπολα είναι μια αρρώστια που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είχαμε και τα επεισόδια στο Forest Area απέναντι σε εθελοντές, τα οποία δυστυχώς ήταν τραγικά επεισόδια, που σημαίνει στη Γουινέα θέλουμε πολύ πιο εξειδικευμένη προσέγγιση του θέματος. τα περιστατικά μέχρι τώρα δεν αυξάνονται όπως στη Σιέρα Λιόνε, αλλά προσωπικά έχω μια έντονη επιφύλαξη το τι συμβαίνει πραγματικά επί του εδάφους. Και αυτό λέγεται και από τους επιδημιολόγους. Είναι γι' αυτό που ζητά και η κυβέρνηση και ήταν καλή συνεργασία, είχαμε μια ειδική συνάντηση με όλους τους υπουργούς και τον National Coordinator χρειάζεται, χρειάζονται ειδικοί επιδημιολόγοι για να μπορέσουν με στατιστικά στοιχεία, με συγκεκριμένα data, να εκτιμήσουν τις περιοχές που πρέπει να στείλουμε τα, ε, ε, ε, να στείλουμε τα treatment centers και να δημιουργήσουμε τα community centers. Η Γουινέα θέλει ειδική επικοινωνιακή communication στρατηγική. Ακόμα και ο πρόεδρος ο ίδιος στη συνάντηση μας το είπε ως κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ίδια την πρωτεύουσα των Κονάκρη υπάρχουν περιοχές που αντιστέκονται να δεχτούν ότι ο έπολα είναι μια αρρώστια που χρειάζεται ιατρική προσέγγιση πιστεύουν ότι είναι κάτι διαβολικό, ότι υπάρχει ένα σε αυτού του ανθρώπου σαν κοσπίραση theory και γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση από τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνα. Κάπου μάλιστα ένας από UN agency μας είπε ότι στην προσπάθεια να επικοινωνήσουν βρήκαν αντίσταση διότι πιστεύουν ότι είναι δυτικός δάχτυλος ε, από ε, την Δύση και ο έμπολα δεν υπάρχει, απλώς όλα αυτά λέγονται για να μπορέσει η Δύση να επιβληθεί στη Γουινέα. Εκεί τα συγκεκριμένα άτομα από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις Μα ζήτησαν όντω ότι χρειάζονται γαλλόφωνοι γαλλόφωνοι επιδημιολόγοι, γαλλόφωνοι άνθρωποι που να ασχοληθούν με τα θέματα της επικοινωνίας του communication και εδώ είναι ακριβώς που ήταν πολύ καλό το ότι έγινε η επίσκεψη στην παρουσία της Υπουργού Ανάπτυξης της Γαλλίας είναι μια... Χρειαζόμαστε τη γαλλική παρέμβαση. Είναι η ιστορία της χώρας, είναι η ίδια η γλώσσα η οποία θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή ότι ε, και είναι πολύ καλό ότι έχει αυξήσει πολύ τις προσπάθειες και την παρουσία της πλέον η γαλλική κυβέρνηση μετά από αυτή την επίσκεψη. Είχε γίνει και το άνοιγμα ενός κέντρου 50 κρεβατιών από την Υπουργό με την ενίσχυση και την χρηματοδότηση και τη δική μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πέρασε ως πάρα πολύ καλό μήνυμα για να περιοριστεί το πρόβλημα της επικοινωνίας και της πυθούς απέναντι στους ε, leaders των communities. Θα σας μεταφέρω το πώς σκεφτόμαστε να ενεργήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής και σε συνεργασία με τα Member States. Πρώτον, στο επίπεδο του medical personnel. Χρειαζόμαστε όντως να πείσουμε ότι πρέπει να πάνε περισσότεροι γιατροί και περισσότεροι νοσοκόμοι και νοσοκόμες. Ήδη εστήραμε επιστολή στους Υπουργούς Υγείας με τον συνάδελφο Ικάτης ενδεχομένως να κάνουμε και μια ειδική συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας όλων των κρατών για να γίνει ειδικό promotion σε κάθε χώρα έτσι ώστε ακριβώς να φτάσουμε στο επίπεδο του medical personnel που υπάρχει ανάγκη. Καταγράφουμε σε κάθε χώρα, είμαστε ήδη σε επαφή με τους National Coordinators Λιβερία, Σιέρα Λεόνε τουλάχιστον, έτσι ώστε να ξέρουμε το επίπεδο των γιατρών που χρειάζονται, πόσες νοσοκόμες. Ελπίζουμε να έχουμε την ανταπόκριση στην οποία έχουν δεσμευτεί στις συναντήσεις. Ζητήσαμε ήδη και τη βοήθεια των Αμερικανών στη Λιβερία και των Βρετανών στην Σιέρα Λεόνε. Για, αν δεν έχουμε την ανταπόκριση από τα συγκεκριμένα κυβερνητικά τμήματα, όχι λόγω του δεν θέλουν, αλλά μήπως δεν μπορούν, γιατί υπάρχει μια δυναμία, τουλάχιστον να μας στείλουν ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συγκεκριμένη ειδικότητα, χρειαζόμαστε αυτούς τους χημικούς για τις αναλύσεις, χρειαζόμαστε αυτούς αυτέ τι νοσοκόμε που ξέρουν αυτή τη δουλειά. Γιατί ενδεχομένω θα πρέπει να γίνουν και training center σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα για αυτοί που θα σταλούν να είναι προετοιμασμένοι. Γιατί δεν θα είναι γενικά ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο ή οτιδήποτε ειδικότητα. Πρέπει να είναι εξειδικευμένο με μικρή βέβαια εξειδίκευση μια εβδομάδα 15 μέρε ή σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του ιού είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία με τους Υπουργούς Υγείας στο επίπεδο του medical personnel. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με τον Commissioner Βιτένης Αντρουϊκάτης. Ήδη ξεκινήσαμε διότι πήγαμε μαζί εκεί και είχαμε και τη συνεργασία εκτός της ΕΚΟ και της ΣΑΝΚΟ. DG. Δεύτερο. Χρειάζονται λεφτά ο συνάδελφο πριν πολύ σωστά είπε ότι πρέπει να βρούμε τρόπου να αυξήσουμε την οικονομική ενίσχυση. Υπάρχει ήδη μια πρωτοβουλία για ένα τραγούδι εναντίον του έμπολα. Έχω κάνει κάποιες επαφές για μεγάλες συναυλίες σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που ταυτόχρονα θα δημιουργούν το κλίμα solidarity στην κοινωνία αλλά θα υπάρχει και οικονομική ενίσχυση. Χρειαζόμαστε μεγάλα γεγονότα στην Ευρώπη κατά του έμπολα. Και οι καλλιτέχνε συνήθω σε αυτέ τι περιπτώσει βοηθούν πολύ γιατί έχουν μια άμεση επαφή με τον απλό άνθρωπο, με την κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε με υπουργού εσωτερικών και άλλα τέτοια σύνολα έτσι ώστε να γίνουν μεγάλες συναυλίες σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Το τρίτο έχει σχέση με το πώς θα περιορίσουμε όντως το πρόβλημα του φόβου και της ιστερίας στις δικές μας κοινωνίες. Γιατί ο έμπολα είναι περίπου όπως το AIDS που περάσαμε αυτή την περίοδο της ιστερίας και μετά απεδείχθη ότι είχαμε δίκιο ότι δεν χρειαζόταν ιστορία. Ο ιός μεταδίδεται μόνο με συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνεται πολύ καλό exit control στις τρεις χώρες, στις τέσσερις, εάν συμπεριλάβουμε και το Μάλι. Εκεί βρήκαμε κατανόηση έτσι ώστε να αυξηθούν τα μέτρα του exit control. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το exit control παρά το entry screening. Το οποίο πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα, αλλά είναι πιο σημαντικό να γίνεται εκεί. Γιατί πιστεύω αγράδαντα μετά και που είδαμε την κατάσταση on the ground ότι τον ιό θα τον νικήσουμε εκεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε να έρθει εδώ για να νικηθεί. Εκεί θα τον νικήσουμε. Και μπορούμε να τον νικήσουμε. Τελειώνω λέγοντας τρία πράγματα. Ότι πριν έρθω εδώ ήμουν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Έγινε μια καλή συζήτηση και έγινε αντιληπτό στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε, δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Το 1 billion point 2 που δεσμευτήκαμε, ίσως και πιο πολύ, θα πρέπει όντως να είναι το ποσό που θα πρέπει να δοθεί για τον εναντίον του έμπολα. Δεν πρέπει να κάνει κανείς πίσω από τις δεσμεύσεις του το κάθε member state, ο κάθε οργανισμός. Είπα αυτά που είπα και τώρα ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να εμπλέξουμε τις κοινωνίες στη συλλογή χρημάτων και βρήκα κατανόηση. Είδα μια αποφασιστικότητα στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών ότι ναι, η Ευρώπη όντως μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας Αντιμετώπιση του ιού μαζί με τους άλλους international partners. Θεωρώ ότι όντως υποτιμήθηκε η κατάσταση ως τώρα, κυρίως μέχρι τον Αύγουστο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και η Επίτροπος Κρυσταλίνα είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από την αρχή, αλλά δυστυχώς υπήρχε μια διεθνής υποτίμηση για διάφορους λόγους. Τώρα κάνουμε μια νέα αρχή. Η δική σας βοήθεια είναι πολύ σημαντική ως Επιτροπή. Ουσιαστικά είσαστε το καμπανάκι που θα μας ευαισθητοποιεί όλους, που θα μας κρατά σε εγρήγορση. Και πιστεύω ότι πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει σαφέστατα σε όποιες πρωτοβουλίες γίνονται να συμμετέχετε πρωταγωνιστικά και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε το ρόλο σας και στο Σάμιτ και στο επίπεδο το πρώτο αλλά και στο δεύτερο. Η παρουσία της Επιτροπής αυτής δείχνει ότι οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να είναι παρόντες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ουσιαστικά είναι τμήμα της συμμετοχής των ευρωπαϊκών λαών σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Δεν αποκλείω και μια ειδική ομάδα από την Επιτροπή να κάνει επίσκεψη στην περιοχή. Δεν είμαι σίγουρος για τις διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει όντως πολύ αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Το χρειάζονται. Χρειάζονται αυτή την ηθική στήριξη από εμά. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πάτε. Τελειώνω λέγοντας σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Ό,τι χρειαστεί θα σας ενημερώνω. Θα στέλνω σημειώματα στην πρόεδρο της Επιτροπής έτσι ώστε να είμαστε ουσιαστικά σε καθημερινή επικοινωνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. We must to act now, not tomorrow. Thanks a lot. ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ήταν ε, το ταξίδι αυτό στις χώρες Δυτικής Αυτής πάρα πολύ καρποφόρο. Εντατικά εργαστήκατε, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω, ε, διότι υπάρχουν εκπρόσωποι ΜΚΟ εδώ, επειδή έχετε πείρα στην ε, επιτόπου εργασία. Θα θέλαμε, για αυτό το ήθελα να σας ακούσουμε και να μας ενημερώνετε λοιπόν ε, για την εμπειρία που έχετε επιτόπου και χρειαζόμαστε να, είμαστε, να ε, παγρυπνούμε, όπως είπε ο Βίτροπος και στις γειτονικέ χώρες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σας χρειαζόμαστε, πρέπει να είμαστε σε επαφή. Τελικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Ε, ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πολύ λεπτό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα τώρα να περάσουμε μηνύματα και στις δικές κοινωνίες για να πούμε σε όλους ότι θέλουμε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει, χρειαζόμαστε κονδύλια και συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπιση του προβλήματος. Σας ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε μαζί σας για την περαιτέρω εξέταση του όλου θέματος στο μέλλον.